So, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας για σήμερα της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Καλώς ήρθατε όλοι ή έχετε μπροστά σας ε, μια ημερήσια διάταξη. Υπάρχει κάποια πρόταση να αλλάξουμε κάτι στην ημερήσια διάταξη. Όχι, οπότε μπορούμε να υιοθετήσουμε την ημερησία διάταξη. Το δεύτερο σημείο είναι το η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 25ης Νοεμβρίου και της Δευτέρας και 3 η Δεκεμβρίου του 2019. Εγκρίνονται εκτός αν υπάρχουν αντιρρήσεις από τα μέλη της ε, Επιτροπής αυτής. Σημείο 3. Ανακοινώσεις των συντονιστών ε, της Δευτέρας Δεκεμβρίου. Και εδώ, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μέχρι το τέλος ε, της συνεδρίασης θα θεωρηθούμε ότι έχουν εγκριθεί. Σημείο 4. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Όπως συνήθως ε, μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή. Οπότε καλωσορίζουμε και τους ανθρώπους από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ταλίν και από την Λισαβόνα μέχρι το Γκέτεμποργκ Έχουμε σχεδόν 700 επισκέπτες κατά μέσο όρο καθημερινά. Είναι αρκετοί. Και φυσικά υπάρχει και διερμηνία. Παρακαλούμε να μιλάτε με κανονική ταχύτητα. Και τρίτον, ήθελα να πω ότι ο Μάρκ Γιούτεν θα εγκαταλείψει την Επιτροπή μας, δυστυχώς, ή μάλλον έχει ήδη εγκαταλείψει την Επιτροπή μας από την 1η Ιανουαρίου. θα μεταπηδήσει στη γραμματεία της ΑΦΕΤ. Θα πρέπει... Έτσι έχουμε και μια επαφή μέσα στην ε, ΑΦΕΤ και αυτό είναι καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κάνατε στην Επιτροπή μας και καλή τύχη στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ο νέος συνάδελφος που αναλαμβάνει το ρόλο του στη γραμματεία είναι ο Ντίντερικ Ντεσμέτ. Καλώς ορίσατε και Καλή τύχη ε, για τη δουλειά σας στην Επιτροπή, ό,τι καλύτερο και καλή υπομονή γιατί ε, είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ πολύ. Α, παρόλα αυτά είμαστε και εντάξει άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, οπότε καλή σας τύχη. Πάμε στο σημείο 5. Η ετήσια ανταλλαγή απόψεων με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε εδώ την κυρία Κέρτης, είναι επικεφαλής κλάδου από το τμήμα Νόρμες, ένα τεράστιο τμήμα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Καλώς ορίσατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά έχουμε μια συνεχή συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ε, στο πλαίσιο πολλών εμπορικών συμφωνιών αλλά και στο πλαίσιο του GPS, της παρακολούθησης ε, και άλλων ζητημάτων. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν ε, οι συναλλαγές μας, ε, οι επαφές μας και ειδικότερα συγκεκριμένα όσον αφορά το 2019 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είχε την εκατοστή της επέτειο. Κυρία Κέρτης λοιπόν καλωσορίσατε και σας δίνουμε αμέσως το λόγο για 15 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όπως θα ξέρετε, είμαστε τριμερής οργανισμός όπου εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις αλλά και οι επιχειρήσεις και οι εργαζομένοι. Η Διεθνής Οργάνωση εργασία παίζει κρίσιμο ρόλο. Διασφαλίζει ίσες συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τους κανόνες εργασίας που είναι απαραίτητοι για βιώσιμες εμπορικές συνεργασίες. Η εντολή μας είναι η πρόθεση των προτύπων και η υποστήριξη και εποπτεία της υλοποίησης μέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς ο οργανισμός μας μπαίνει στο δεύτερο αιώνα λειτουργίας του. Με την ευκαιρία θα σας παρουσιάσω τις εξελίξεις που είχαμε πέρυσι ε, κατά την 100 ε, επέτειο του ILO και θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει τη δική σα επιτροπή στο σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Να σα υπενθυμίσω λίγο τα θέματα που οδήγησαν στη δημιουργία του ILO και πόσο σημαντικό ήταν για να δημιουργήσει ένα χώρο, ε, ένα περιβάλλον ε, ισότιμου εμπορίου. Δεν θέλω να θεωρείτε ότι είναι κάτι δεδομένο ο οργανισμός αυτός και η φήμη του. Δεύτερον, θα παρουσιάσω τα πρότυπα και τη ρύθμιση προτύπων και την εποπτεία των προτύπων του ILO που τον κάνουν να αποτελεί σημαντικό ε, σημείο αναφοράς ε, στο διεθνές ε, δίκαιο εργασίας. Επίσης θα σας πω με την ευκαιρία της 100 επαιτίου τους στόχους και τις συνέργειες. Θα σας παρουσιάσω τις χώρες και τα ζητήματα που εποπτεύει. Και τέλος θα ολοκληρώσω Παρουσιάζοντας σα πώ μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιολογούμε και να επιβάλλουμε την, τα πρότυπα ε, με του εταίρου μα στην Ευρώπη. Πρώτον, από την δημιουργία του μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις τάχτες του, ο ILO και η εντολή του δημιούργησε το περιβάλλον για διεθνή εργασιακά πρότυπα ως βασικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες. Ο αθέμητος ανταγωνισμός ως έννοια και ο αγώνας προς τα κάτω οδήγησαν στην δημιουργία του όπου δηλώθηκε ότι η αποτυχία ενός κράτους ε, να εφαρμόσει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αποτελεί εμπόδιο και για τις άλλες χώρες που θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες αυτές. Κατ' επακόλουθο, η δήλωση του 1918 για ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων δέσμευε όλους τους οργανισμούς. Η εκρίζωση της αναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας, η ποιότητα της εργασίας και η ελευθερία ε, του συνεταιρίζεστε και των συλλογικών συμβάσεων. Μία δεκαετία αργότερα η παραβίαση αυτών των θεμελιωδών αρχών δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα πλέον την είχαν υιοθετήσει όλα τα μέρη του ILO στην δήλωση για την κοινωνική δικαιοσύνη και δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό το σκοπό η δήλωση δημιούργησε χώρο για τον ILO να παρέχει αρρωγή στα μέλη που ήθελαν να προωθήσουν τους στόχους του από κοινού στο πλαίσιο δημερών ή πολυμερών συμφωνιών. Αυτό με οδηγεί στο δεύτερο μου σημείο που αφορά τη σπουδαιότητα των προτύπων και της εποπτείας του ΑΕΛΟ ως εργαλείων εμπορικών. Ο ΕΛΟ απέκτησε την ομοποίησή του ω σημείο αναφορά στον τομέα τη εργασία λόγω των μηχανισμών που χρησιμοποιεί χωρί αποκλεισμού, οι οποίοι ρυθμίζουν πρότυπα για διάλογο βάσει συνένεση με την παγκόσμια κοινότητα, τη επιχειρήση και του εργαζομένου. Είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο σύστημα εποπτείας που συνδυάζει υποβολή αναφορών και αξιολόγηση βάσει καταγγελιών, ε, πολυμερών και βάσει αξιολόγηση Ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης ε, καθιστά τον ΑΕΛΟ απαράμιλο ως θεμέλιο ε, συγκριτικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Τρίτον, δεδομένης της εκατοστής επαιτίου, δεν μας εκπλήσει ότι η επέτειος αυτή μας κάνει να θυμηθούμε τα επιτεύγματα που χρήζει να υπογραμμίσουμε σήμερα που συνεχίζουν να είναι πολύ σημαντικά και καθορίζουν την σπουδαιότητα του ILO ως οργανισμού καθορισμού προτύπων. Πρώτο-πρώτο με τεράστια υποστήριξη, όπως βλέπουμε στην ετήσια διάσκεψη για την εργασία για την υιοθέτηση της συνθήκης 190 του ILO για ένα σημαντικό θέμα για τον κόσμο εργασίας σήμερα είναι η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη στη διάσταση του φύλου παρέχει το πλαίσιο που αναμένει η διεθνή κοινότητα ούτως ώστε να προλαμβάνεται και να ε, επανορθώνεται η βία και η παρενόχληση στον χώρο της εργασίας. Η Τριμερής Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων έκανε εντατικέ συζητήσει για την παγκόσμια έρευνα που έγινε από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων βάσει μια πρόσφατα υιοθετημένη σύσταση για την κοινωνική προστασία. Αναδείχθηκε η σπουδαιότητα τη κοινωνική προστασία στην παγκόσμια αναπτυξία Γκέντζαδα και πόσο σημαντική είναι η σύσταση για να καθοδηγήσει τη δράση καταπολέμηση τη φτώχεια, τη ανισότητα, τη κοινωνικού αποκλεισμού και για να επιτευχθούν παγκόσμια δικαιώματα που διασφαλίζουν αξιοπρεπή υγεία και ζωή. Ε, το άλλο βασικό καθήκον τη Επιτροπή Εφαρμογή είναι να επιλέγει και να συζητά 24 υποθέσει που αφορούν την εφαρμογή ε, επικυρωμένων ε, συμβάσεων που πρέπει να εξετάζονται τριμερώς. Όπως θα αναμενόταν, πολλές από αυτές τις υποθέσεις αναφέρονται σε σημαντικά προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή βασικών η εφαρμογή τη ελευθερία του συνεταιρίζεστε και της ε, συλλογικής, των συλλογικών συμβάσεων είχε υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα. Έγιναν συζητήσεις για την Αλγερία, τη Βραζιλία, την Αίγυπτο, τα νησιά Φίτζη, την Ονδούρα, το Καζακστάν, τις Φιλιππίνες, την Ουρουάη και τη Ζιμπάμπουε. Η περίπτωση του Καζακστάν επισημάνθηκε ως ιδιαίτερη Εκεί παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις υλοποίησης της ε, ε, επικυρωμένη σύμβάση. Ε, οι περιπτώσει παιδική εργασία αφορούν το Πράσινο Κροτήρι, την Αιθιοπία, το Ιράκ και το Λάο, Ενώ έγιναν συζητήσει για την κατάσταση τη αναγκαστικής Εργασία στη Λευκορωσία και στη Μιαμάρ. Η Λαβή και το Τατζικιστάν επίση συζητήθηκαν όσον αφορά τη συνθήκη για τη διακριτική μεταχείριση στον χώρο εργασία οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι τριμερείς διάλογοι έχουν ειδική θέση ως πρότυπα στον ILO και σχετίζονται με αυτό που παρατηρούμε στην Ινδία και στη Σερβία για την επιθεώρηση εργασία και με το Σαλβαδόρ για το δεύτερο θέμα για την τριμερή διαβούλευση. Τέλο, Τέλος, οι συζητήσεις για τις τεχνικές συνθήκες συμπεριλαμβάνουν τη Βολιβία ε, και την Ικαράγουα σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Συμπεράσματα που έχουν συμφωνηθεί με συνένεση και με συστάσεις για δράση γίνονται για κάθε συζήτηση. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αλλά θα σας προσθέσω στα βασικά σημεία. Η Βραζιλία είναι μια περίπτωση όπου βλέπουμε το σημαντικό ζήτημα ε, και τους σκοπούς των συλλογικών συμβάσεων. Το 2017 υποβλήθηκαν νομοθετικές ε, ε, τροπολογίες που δίνουν τη δυνατότητα στις συμβάσεις να παρεκκλίνουν από την νομοθεσία με εξαίρεση τα δικαιώματα που υπάρχουν στο Βραζιλιανικό Σύνταγμα. Στην, Επιτροπή, στην Τριμερή Επιτροπή θεωρήθηκε ότι δεν πληρείται εδώ οι συνθήκες για την πρόθεση των συλλογικών συμβάσεων και έγινε σύσταση να εξετάζονται οι επιπτώσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή Εμπρογνωμόνων θεώρησε ότι ενώ οι συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν συγκεκριμένες διατάξεις, συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας ε, μπορούν να αιτιολογήσουν ε, περιορισμένες εξαιρέσεις ε, και είναι συμβατές με τη συνθήκη μια γενική διάταξη που προβλέπει ε, την εξαίρεση κάποιων διατάξεων προστασίας της εργασίας έρχονται σε αντίθεση με τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την ιεραρχία της νομοθεσίας, όπου η νομοθεσία γενικά θεωρείται ότι υλοποιείται ως ελάχιστο πρότυπο και οι συλλογικές συμβάσεις απλά παρέχουν καλύτερες συνθήκες όπου είναι δυνατόν για τους εργαζομένους. Στην περίπτωση της Αιθιοπίας, η τριμερή συνάντηση θεώρησε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για την γενική επιθεώρηση, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα ανθρωπιστικά και οικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε να μην υπάρχει καταναγκαστική εργασία στην Αιθιοπία. Επειδή ε, υπάρχει και το θέμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να μην υπάρχει εργασία ανηλίκων, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να επιβληθεί μέχρι τα 14. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γενική διακήρυξη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας το 2019 σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Επίσης, στην Ινδία έγιναν συστάσεις με στα πλαίσια της Γενικής Επιτροπής Επιθεώρησης, έτσι ώστε οι επιθεωρητές να μπορούν να κάνουν και ε, ε, απρόοπτες ε, μη προγραμματισμένες αυτοψίες, λαμβάνοντας υπόψη και την συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε και η αυτοεπιθεώρηση να μην συρρυκνώσει τη, τις αρμοδιότητες του ΔΟΕ. Στο Μιανμάρ λαμβάνουμε υπόψη την συνέχεια των συστάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής που συστάθηκε το 2019. Η Τριμερής Επιτροπή ζήτησε από την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμβάσεις από πλευράς στρατιωτικών ή πολιτών και ακριβώς για να μην υπάρχει εκμετάλλευση και εργασία ανηλίκων. Αυτό αφορά και μία μετάβαση ε, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε και τα παράπονα που υπάρχουν στον τομέα της ε, υποχρεωτικής εργασίας ανηλίκων. Στην, ε, στις Φιλιππίνες είδαμε το θέμα της ατιμορρησίας στον τομέα της εργασίας και την βία κατά των συνδικάτων. Η Τριμερής Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα και κυρώσεις έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα και καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Επίσης, θα πρέπει να συσταθεί μία Τριμερής Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται αυτό το πλαίσιο. Ο ΔΟΕ επίσης έχει προωθήσει ε, έναν μηχανισμό κύρωσης μέσα στα πλαίσια της πανηγυρικής επαιτίου των 100 χρόνων. Επίσης, ασχολείται με την αναθεώρηση των ε, συνθήκων εργασίας για να είναι εύρωστες και δίκες. Με την ενίσχυση αυτών των μηχανισμών, ο ΔΟΕ, ανά τις δεκαετίες αυτές, προώθησε την σωστή εφαρμογή των συμβάσεων. Οι θεμελιώδεις συμβάσεις του ΔΟΕ έχουν τονίσει ιδιαίτερα τις συνέργειες μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων έτσι ώστε να φτάσουμε σε κοινού στόχους. Το ε, τμήμα των προδιαγραφών του ΔΟΕ προωθεί το θέμα της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα εργασιακά δικαιώματα. Με την υποστήριξη της ΔΕΒΚΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου προβήκαμε σε καλύτερα, καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου στο Κάμπο Βέρτε, Αρμενία, Μογγολία, Μιανμάρ, Πακιστάν, Παραγουάι, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ για την αξιοπρεπή εργασία προωθούμε αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να προβούμε σε μια συγκεκριμένη στοχοθέτηση κρατών. Όχι μόνο για να ε, δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά και για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς εμπορικές προδιαγραφές. Προδιαγραφές διεθνούς εμπορίου. Παρά το γεγονός ότι στις Φιλιππίνες πίνες ε, υπάρχει μία απόκληση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τα όργανα αντιμετώπισης της ατιμορρησίας στις, στις Φιλιππίνες. Η διακήρυξη των 100 ε, ετών ορίζει και τις ε, πολυσχηδείς προκλήσεις αυτών των τελευταίων ετών μετά την παγκοσμιοποίηση. Έτσι προβήκαμε στην χαρτογράφηση των προτεραιοτήτων όσο προχωρούμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εμπορικές πολιτικές για να υπάρχει προβλεψιμότητα. Πέρσι το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε συγκεκριμένες συστάσεις και αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των ε, συνθήκων εργασίας για να μην υπάρχει ατιμορρησία και να μην υπάρχει και ανισότητα στους όρους εργασίας. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με τη δική σας Επιτροπή αφορούν μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στο πολύπλευρο εμπορικό πλαίσιο και αυτό αφορά και τις βιομηχανικές πολιτικές. Η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη εξαρτάται από αυτή τη συνοχή και χαίρομαι που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συγκεφαλαίωση. Και θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας, ξεκινώντας κυρία Βαγιά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Υποστηρίζουμε το έργο σας, τις προσπάθειές σας. Έχω ένα ερώτημα σε σχέση με το κατά πόσο πιστεύετε ότι εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, τα πρότυπα αυτά, στις Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικότερη και καλύτερη εφαρμογή των ε, διατάξεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ε, για την γενική και πλήρη παρουσίασή σας του έργου του ΔΟΕ. Θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για τις διμερείς συμφωνίες Συνεργαστέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Είπατε στην παρουσίασή σα ότι αυτέ έχουν θετικά αποτελέσματα. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω το εξή. Πώ συνεργάζεστε πιο συγκεκριμένα με την Επιτροπή, αλλά πιθανώ και με άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχει παρακολούθηση των λεγόμενων κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχουμε σε αυτέ τι συμφωνίε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Μας δώσετε μια γενική εικόνα, πολύ σημαντική. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι πιο γενική. Ε, πέρα από συγκεκριμένες χώρες τις οποίες εξετάσατε, μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση θετική ή αρνητική στο κατά πόσον εφαρμόζονται οι συμβάσεις του ΔΟΕ. Και κάτι που πιο συγκεκριμένα αφορά και την Επιτροπή μας. Τι διαπιστώνετε όταν υπάρχει μια εμπορική σχέση, είτε με ελεύθερη συμφωνία εμπορίου, είτε με GSP, είτε με κάποιο τέτοιο είδους πλαίσιο. Βλέπετε να, να δημιουργείται θετικός αντίκτυπος, βοηθάει. Και όπως και οι άλλοι συνάδελφοί μου θα ήθελα να μου πείτε σε σχέση με άλλα πρότυπα, μάλλον σε σχέση κυρίω με τα πρότυπα τα οποία αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οποία βασίζονται ε, κυρίω στην επιβολή κυρώσεων. Πώ πιστεύετε ότι μπορούμε να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε πιο αποτελεσματικά. και στον τομέα των ενδιαφερόντων των δικό σα, δηλαδή του ΔΟΕ ή και σε άλλου τομεί, Πιστεύετε ότι πρέπει να αρχίσουν να δημιουργούνται νέα διεθνή πρότυπα, χρειαζόμαστε νέα διεθνή πρότυπα. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Κύριε Χάουτελα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γνωστό, είναι αυτοπόδεικτο, είναι προφανές ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι ένα σημαντικό εταίρος τη επιτροπή μας. Ε, πολύ συχνά είναι, αποτελούν εμπόδιο για τις ε, συμφωνίες ελευθέρων εμπορίου ή συνθήκε εργασίας σε μια χώρα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι το οποίο συνδέεται και με την ψηφοφορία που θα έχουμε αύριο για τη Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου με το Βιετνάμ. Αν και διαπιστώσαμε ότι το δίκαιο, το εργατικό σε αυτή τη χώρα βελτιώνεται, θα πρέπει να το εξετάσουμε σε σχέση με τα πισωγυρίσματα που έχουμε διαπιστώσει στον ποινικό κώδικα. Για παράδειγμα, μπορεί στο, εργατικό δίκαιο να αναγνωρίζεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, όμως αυτό το δικαίωμα μπορεί να ε, εξουδετερώνεται από άλλες διατάξεις που μπορεί να υπάρχουν στον ποινικό κώδικο. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Θα γνωρίζετε ότι σε πολλές πολιτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου συζητούμε τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δέουσας επιμέλειας για την προστασία αυτών. Έχουμε διαπιστώσει πολλά ενισχυτικά περιστατικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για χώρες όπως για παράδειγμα η Μαλαισία που είναι ένα σημαντικός ε, παραγωγός ε, καουτσούκ ε, ελαστικών προϊόντων στον κόσμο. Και διαπιστώνουμε καταχρήσεις και εξαναγκαστική εργασία μέχρι και σκλαβιά θα μπορούσε να ονομάσει την κατάσταση κανείς. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αντιμετωπίζει κανείς μια τέτοια κατάσταση Ιδίω δεδομένου ότι ήδη από το 2016, αν δεν απατώμε, έχει επιβληθεί ένα εμπάργκο σε προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με καταναγκαστική εργασία σε, σε, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αυτό το καταλληλότερο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των εργαζομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι οι κοινωνίες μας έχουν μηδενική ανοχή στην εξαναγκαστική εργασία, στη σκλαβιά. Πώς αντιμετωπίζει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας τέτοιες περιπτώσεις και τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές κατά την απόψή σας. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Το δικό μου ερώτημα συζητείτε, έχει σχέση μάλλον με μια άλλη συμφωνία ελευθερών πορείου που θα συζητήσει η Επιτροπή μας. Αναφερθήκατε στη Βραζιλία. Και αν, δεν, αν σας κατάλαβα κατά, είπατε ότι δύο επιτροπές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας είχαν διαφορετική αξιολόγηση της κατάστασης εκεί. Θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα τι κάνει ο ΔΟΕ για να αντιμετωπίσει την προσπάθεια του Προέδρου Μπολσονάρου να καταστρέψει το εργατικό δίκαιο στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Είναι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη που άργησα να έρθω, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και γενικότερα να σας συγχαρώ για τον εξαιρετικό έργο του ΔΟΕ. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Πώς αξιολογείται το, την έκθεση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής για το κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε πλέον στις συμφωνίες ελευθερών εμπορίου και πώς θεωρείτε ότι αυτό μπορούμε να το ενισχύσουμε και να το εμβαθύνουμε. Δεύτερον, σε χώρες που έχουμε ένα αναπτυγμένο αργατικό δίκαιο που διαπιστώνεται όμως ότι υπάρχει ένα, μια υποστοχώρηση Ποια είναι η δική σας η αξιολόγηση. Ε, για παράδειγμα, έχει κάποιες ε, επικριτικές συστάσεις να απευθύνει ο ΔΟΕ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χώρες οι οποίες τις θεωρούμε συνήθως ανεπτυγμένες από πλευράς εργατικού δικαίου. Ιδίω, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου έχουμε υποβάθμιση των εργατικών προτύπων εξαιτία της οικονομικής κρίσης, κάτι που διαπιστώσαμε να συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης. και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προωθήσουμε συστήματα τα οποία να προβλέπουν ακυρώσει έτσι ώστε να ε, υπάρχει ουσιαστική εφαρμογή των διαφόρων δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις σε θέματα εργατικού δικαίου, εργατικών συνθήκων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και με έναν ε, από στους συναδέλφους σας στο παρελθόν. Ε, είπατε ότι υπήρξε μια μεγάλη επιτάχυνση στην εφαρμογή των συμβάσεων του ΔΟΕ ε, από τη στιγμή που ξεκινούν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπεριλαμβάνουν και τέτοιο σχετικό κεφάλαιο. Το βλέπουμε αυτό, θα το συζητήσουμε και στη συζήτησή μας αύριο για το Βιετνάμ. Έχουμε δημιουργήσει την ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου μα από το Βιετνάμ, εμεί οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το πώ θα, ε, ε, εφαρμόσουμε αυτό το, αυτή την προσπάθεια, αυτό το θεματολόγιο. Θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία με το Βιετνάμ θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα, πρότυπο για μελλοντικέ μα συμφωνίε με τρίτε χώρε. Και αν ναι, τι πιστεύετε ότι είναι το ιδιαίτερο στοιχείο που προσέθεσε αυτό το εργαλείο. Ευχαριστώ. Δύο ε, πράγματα να προσθέσω. Συμφωνώ με πολλές από τις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Εμείς ως Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου δεν είμαστε μόνο αρμόδιοι για αποφάσεις που αφορούν το εμπορίο, αλλά και για την εφαρμογή. Θέλουμε να βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται στην πραγματικότητα για τα ζητήματα αυτά, για το βιώσιμο κεφάλαιο, για την πολιτική απασχόληση, για σημαντικέ πολιτικές. Οπότε εγώ θα ήθελα να μάθω εσείς ως ILO, ως ΔΟΕ, ε, πώς εκτιμάτε, πώς ε, ε, παρακολουθείτε το ζήτημα, πώς να το πω, της υλοποίησης. Δηλαδή κάνετε κάτι, έχετε domestic advisory groups, τι γίνεται όσον αφορά την παγίωση των εργασιακών προτύπων. Στην πραγματικότητα, κατά την άποψή σας, τι πρέπει να λαμβάνουμε εμείς ε, όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για νέες συμφωνίες. Τι πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο. Εκεί τίθεται το ερώτημα. Δηλαδή, ποιε διαδικασίε, πώ ε, γίνονται τέτοιοι μηχανισμοί δηλαδή αξιολόγηση, του οποίου χρειαζόμαστε, τι θα χρειαστούμε σε 10 χρόνια από τώρα. Ε, τι πρέπει να κάνουμε για να δούμε τι έχει βελτιωθεί πραγματικά και τι όχι. Ούτω ώστε να βελτιώσουμε και την οικονομική συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των κρατών μελών και των τρίτων χωρών αλλά και εντός των ίδιων περιοχών, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δεύτερη ερώτηση που θα με ενδιαφέρε. Έγινε μια διάσκεψη για τη συμφωνία ε, με την Μερκοσούρ και εμείς ως ομάδα ε, θεωρούμε ότι η Βραζιλία βρίσκεται σε πολύ κακή θέση. Ανεξαρτήτως ε, των συμφωνιών που έχουμε στην εμπορική πολιτική, η νομοθέτηση στη Βραζιλία ουσιαστικά είναι αυθαίρετη. Μπορεί η αστυνομία να κάνει ό,τι θέλει. Ουσιαστικά ατιμόρυτη μπορεί να αποκλίνει από τα πραγματικά γεγονότα, να χρησιμοποιεί όπλα, ε, πυροβόλα, να απειλήσει ε, ζωές ε, ατιμόρυτα, χωρίς καμία συνέπεια και πιστεύω ότι τέτοιες ε, πτυχές ε, της κοινωνικής πραγματικότητας σε τέτοιες χώρες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, στην εμπορική πολιτική. Οπότε και εμείς καλούμαστε να δράσουμε για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πραγματικές συνθήκες σε αυτές τις χώρες. Θέλω να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσε αυτό να αποτυπώνεται σε αυτά τα πρότυπα, σε αυτή την νομοθέτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέρτης. Αναφέρεται την κατάσταση στο Καζακστάν. Το Καζακστάν θα, θα φιλοξενήσει μια τεράστια εκδήλωση του MC τον Ιούνιο και θα πάνε πολλές αντιπροσωπείες. Η, η, πολιτική, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα πάει στο Καζακστάν. Οπότε εκεί ίσως να έχουμε κάποιο πλεονέκτημα στη συζήτηση με την κυβέρνηση του Καζακστάν. Τι θα μας συμβουλεύατε. σε τι θα πρέπει πρωτίστως να εστιαστούμε στη συζήτησή μας για βελτίωση της κατάστασης ε, βάσει των ε, συνθήκων της ε, ΔΟΕ. Πολλές ερωτήσεις και έχετε τώρα εσείς το λόγο για να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω στο μέτρο του δυνατού και θα ήθελα να με επαναφέρετε στην τάξη αν παραλείψω κάτι. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις γενικότερης υφής και πώς ο ΔΟΕ ερμηνεύει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το εμπορικό δίκαιο και θα ε, επισέλθω και σε ορισμένα ειδικότερα ζητήματα. Ο ΔΟΕ, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, δεν είναι κυρωτικό όργανο. Στο Μιανμάρ βέβαια προσπάθησε να το κάνει ιδιαίτερα σε σχέση με την εργασία ανηλίκων που ισχύει από τις αρχές του αιώνα. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις έμπρακτα προσπαθεί να ορίσει ένα γενικό πλαίσιο εργασίας και προδιαγραφών σε σχέση με επιτόπιες καταστάσεις. Και αυτό γίνεται μέσω διαλόγου, άρα προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο διάλογο με την κυβέρνηση και στα πλαίσια και του κοινωνικού διαλόγου σε συγκεκριμένες χώρες. Και οι συμφωνίες σχετίζονται από τη μία πλευρά με τους μηχανισμούς έτσι ώστε να υπάρχουν ομάδες εσωτερικού ελέγχου και ένα πλαίσιο σωστής, σωστών εργασιακών προδιαγραφών. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές και στα πλαίσια των δικών μας οργάνων επιθεώρησης, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή των προδιαγραφών του ΔΟΕ στις χώρες, δηλαδή ως προς τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συμβάσεις του ΔΟΕ που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εμπορικές συμφωνίες. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη δέσμευση στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, συνεργασίας μας, διότι μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε από κοινού τις ε, κατά προτεραιότητα χώρες όπου χρειάζεται δράση αλλά και ένα άνοιγμα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση επιτοπίως και να ορίσουμε τους τομείς που άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων, δηλαδή του ΔΟΕ. Μπορέσαμε λοιπόν να ορίσουμε προγράμματα δράσης και χαρτογραφήσεις για να γίνουν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση με το Βιετνάμ υπήρξε πίεση ως προς την εμπορική συμφωνία για το ΔΟΕ. Η κύρωση μιας συμφωνίας είναι ένα κρίσιμο βήμα. Δεν φαίνεται τόσο σημαντικό, αλλά έτσι εξασφαλίζουμε τη συνεχή αναθεώρηση και εφαρμογή των μηχανισμών του ΔΟΕ. Χωρίς λοιπόν την κύρωση δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα. Γι' αυτό η κύρωση είναι, το κυρωτικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια και η ίδια η εφαρμογή των οδικών χαρτών που δέχονται οι κυβερνήσεις λόγω πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή εμείς στυλιτεύσαμε συγκεκριμένες ε, πολιτικές. Έτσι επιτύχαμε πολλά. Ως προς το Βιετνάμ έγινε λόγος για τον ε, εργατικό κώδικα και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα άνοιγμα ως προς το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε στις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ΔΟΕ, γιατί θα μπορέσουμε να συνοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία τη στιγμή που έχει κυρωθεί αυτό το πλαίσιο. Αυτό αφορά και τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις Εστιάζετε λοιπόν την δική σας προσοχή στις εμπορικές συμφωνίες και εμείς στον μηχανισμό ελέγχου. Έτσι, τα γραφεία μας που βρίσκονται επί τόπου μπορούν να ελέγχουν το πλαίσιο εφαρμογής και να υπάρχει και μια σωστή μόχλευση έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει και μια ενδυνάμει χρήση του ποινικού δικαίου εκεί που υπάρχουν παραβάσεις. Έτσι, η νομοθεσία να συμβαδίζει με τις συμβάσεις του ΔΟΕ στις χώρες αυτές. Αν δούμε το γενικότερο πλαίσιο και τις τάσεις που διαγράφονται, δεν ήθελα να πω πόσο καιρό έχω δουλέψει στο ΔΟΕ, αλλά έχω δουλέψει σε διεθνείς οργανισμούς εδώ και 32 χρόνια. Και συμμετείχα και σε, αυτή, σε αυτόν τον πανηγυρικό εορτασμό του ΔΟΕ. Μιλάμε λοιπόν για διεθνείς συμφωνίες εργασίας, για συλλογικές συμβάσεις, για εμπορικές συμφωνίες. Όλα αυτά είχαν μεγάλη σημασία για την ε, διαδικασία μόχλευσης και για να μπορέσει ο ΔΟΕ να βοηθήσει και να επιβληθεί σε χώρες που δεν μπορούσε διαφορετικά. Υπήρξε και ένα ζήτημα της αιτιόδου συνάφειας με τους ε, ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ΔΟΕ χαίρεται διότι είναι ο θεματοφύλακας συγκεκριμένων δικτών και στόχων μέσα στα πλαίσια ε, αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα από τα θέματα αυτά είναι οι συλλογικές συμβάσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας. Είμαστε θεματοφύλακες αυτού του πλαισίου και χρησιμοποιούνται οι αποτιμήσεις του Μηχανισμού Επιθεώρησης και Ελέγχου του ΔΟΕ για να δούμε ποσοτικά κατά πόσο έχει επιτευχθεί πρόοδος ως προς τις ε, συλλογικές συμβάσεις και το δικαίωμα του συνέρχεστε. Αυτό αφορά και άλλες εμπορικές ε, συμφωνίες και διευθετήσεις για να δούμε αν υπάρχει ε, παλινδρόμηση ή όχι. Επίσης ε, υπάρχει και το θέμα της ίσης αμοιβή για ίση εργασία και αυτό μας δίνει ένα επιπρόσθετο πλαίσιο ε, διακριτικής ευχέρειας και παρέμβασης. Εμείς είμαστε μια τριμερής ε, οργάνωση και γι' αυτό ακριβώς το οποιοδήποτε σκέλος της οργάνωσης μπορεί να έρθει στο προσκήνιο και να μας πει κατά πόσο δεν εφαρμόζονται οι συμβάσεις σε επιτόπια. Αυτό συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ετέθη το ζήτημα της Βραζιλίας στη Συμφωνία Μερκοσούρ, για παράδειγμα. Θα ήθελα να διασαφηνίσω καταρχήν ότι υπήρξαν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε σχέση με τις συλλογικέ συμβάσεις και τις διαπραγματεύσεις για αυτές. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια είναι η θέση της ε, Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που θεωρεί ότι υπάρχει ουσιώδες πρόβλημα τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται η εφαρμογή του δικαίου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγών κατά της κυβέρνησης. Στην περίπτωση της Βραζιλίας ίσχυσε στη, από ε, ομάδες των ε, πολιτών σε σχέση με την σύμβαση ως προς την ε, αντιμετώπιση των αυτοχθόνων. Έχει συσταθεί λοιπόν ένα σώμα για να εξετάσει την κατάσταση και να προβεί σε συστάσεις. Αυτά μέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου με την κυβέρνηση γιατί θέλουμε να προβούμε σε συστάσεις, να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και να δούμε ποια είναι τα κένα και τι δυνατότητα μόχλευσης υπάρχει. Θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη λήψης δράσης από τις κυβέρνησεις ως προς τις συστάσεις. Ως προς τις νέες μορφές εργασίας, τη νέα τυπολογία εργασίας και κατά πόσο χρειάζονται νέες προδιαγραφές, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα συντάξει μία έκθεση που θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο. Μιλάμε για οκτώ μέσα και συνιστώσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα της νέας τυπολογίας εργασίας γιατί υπάρχουν συστάσεις ως προς τη σχέση εργασίας, ε, ως προς την κατοίκο απασχόληση, για παράδειγμα, και πώς αυτά συνδέονται. Θέλουμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο υπάρχουν επιπτώσεις σε σχέση με την απασχόληση και τις σχέσεις απασχόλησης και κατά πόσο υπάρχει μια σωστή παραγωγική απασχόληση. Από αυτή την έκθεση που θα συζητηθεί στη Διεθνή ε, Σύσκεψη Εργασίας θα δούμε κατά πόσο τα μέλη του ΔΟΕ θα ζητήσουν να υπάρξουν νέες προδιαγραφές στο μέλλον. Αυτό θα το δουν τα μέλη του ΔΟΕ εν καιρό. Ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, συγκεκριμένη δράση ως προς την καταναγκαστική εργασία και ούτω καθεξής και τη δέουσα επιμέλεια, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φτάσουμε στην ε, επιχειρηματική κοινωνία ε, και αυτό αφορά σε εθνικό και μη επίπεδο για να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες σε σχέση με την ε, τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας. Αυτό μας επιτρέπει να μπορέσουμε να μιλήσουμε στις, με τις εθνικές οργανώσεις, τις επιχειρήσεις, αλλά και στις, και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως προς το Καζακστάν, Τονίστηκε ιδιαίτερα η περίπτωσή του, γιατί υπήρξε, υπήρξαν σοβαρές παραβάσεις και αδυναμίες σε σχέση με το δικαίωμα του συνέρχεστε, είτε πρόκειται για συνδικάτα, είτε οργανώσεις, οργανώσεις επιχειρηματιών και εργοδοτών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί εάν δεν υπάρχει σωστή εκπροσώπηση, σε επίπεδο συγκεκριμένες χώρας, τότε αποδυναμώνεται η ίδια η οργάνωση. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε ε, αναλάβει μία αποστολή σε τριμερές επίπεδο εδώ και δύο χρόνια, όπου συντάχθηκε ένας οδικός χάρτης για να τροποποιηθεί η νομοθεσία και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να συμμετέχουν στα συνδικάτα που επιθυμούν και αυτό αφορούσε και τους ε, εργοδότες για να υπάρχει ένας ε, κοινωνικός διάλογος ουσίας στη χώρα. Δυστυχώς ε, δεν υπήρξε πρόοδος. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία, οι προδιαγραφές, τα προσχέδια νόμου, αλλά αυτοί οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμοστούν κατ' και υπό το πνεύμα των αλλαγών που έχουν ε, θεσπιστεί. Αλλά επειδή θέλουμε να τονίσουμε στην κυβέρνηση τη σημασία της εφαρμογής και της κύρωσης αυτού του πλαισίου για να ανοίξουμε την πόρτα στο δικαίωμα του συνέρχεσε του συνέρχεστε σε αυτή τη χώρα, το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας. Η κυβέρνηση Νομίζω ότι έχει αρχίσει να αισθάνεται την εξωτερική πίεση. Θα προσπαθήσουν να εργαστούν εντάχει στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και το θέμα δεν θα είναι και ιδιαίτερα ε, προβληματικό τη στιγμή που υπάρχει πολιτική θέληση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, Είμαι σίγουρη αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Εάν ε, παρέλειψα κάποιον, παρακαλώ να μου το πείτε, δευτερολογήσει και ευχαριστώ να απαντήσω. Πρόεδρος, θα έλεγα ότι στο περιεχόμενο, στην ουσία των ερωτήσεων απαντήσατε συνολικά. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα στην κυρία Μαντλέν Τούνιγκα, που είναι υπεύθυνη του τμήματος ε, για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Εργαζόμαστε από κοινού στην ε, Γενική Διεύθυνση Trade και στη Γενική Διεύθυνση Employment ε, εργασία για το ζήτημα αυτό. Επομένω, με την άδειά σα, κύριε Πρόεδρε, να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Πράτ από τη Γενική Διεύθυνση Εργασία. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ει βάθο τι εργασίε του Διεθνού Οργανισμού ε, Εργασία και συνεργαζόμαστε τακτικά. Υπάρχει πολύ ε, καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη στη Γενέβη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με ενιαία φωνή στο ΔΟΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για να ασκηθεί ε, οξία κριτική σε κάποια χώρα για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου ή των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ωστόσο, καταφέρνουμε να έχουμε μια πολύ ε, ε, συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην προηγούμενη διάσκεψη του ΔΕΟ που συζητήθηκε ένα νέο διεθνές πρότυπο και επίσης για την επικύρωση της ε, συμφωνία, του Συμφώνου 119 για την παρενόχληση στον χώρο εργασία. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Και αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υποστηρίζει τι πολυμερεί διαπραγματεύσει, που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και υπ' αυτή την έννοια οι προτεραιότητε αυτών των δύο οργανισμών ταιριάζουν. Έχει δύο σημαντικούς ρόλους να παίξει εδώ. Ε, πρώτα απ' όλα είναι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων ε, και αυτό έχει συμβεί ιστορικά, αν το δει κανεί, από την ίδρυσή του. Το 1920 είχαμε το πρώτο πρότυπο για την ε, εργασία στη θάλασσα, για τους ναύτες. Αργότερα αντίστοιχα πρότυπα για την αλληλεία με ε, ζητήματα που, που ρυθμίστηκαν σε σχέση με τις αμοιβέ των αλλιέων ή για το χρόνο ανάπαυσής τους ή για τον τρόπο αμοιβή τους. Και το δεύτερο, ο δεύτερος σημαντικός ρόλος του ΔΟΑ είναι η παρακολούθηση αυτών των προτύπων και η εντοπισμό των παραβιάσεων. Όλα αυτά πρότυπα αυτά είναι διεθνή πρότυπα. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια επιβολή συγκεκριμένων προτύπων ή συγκεκριμένων απόψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τρίτες χώρες. Πρόκειται για διεθνή πρότυπα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ΔΟΕ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του ΔΟΕ είναι ακριβώ ότι υπάρχει η τριμερή διαπραγμάτευση, ότι υπάρχει εκπροσώπηση και των κυβερνήσεων και των εργαζομένων και των εργοδοτών με του αντίστοιχου εμπειρογνώμονε. Ε, και αυτό όχι μόνο επειδή υπάρχει εκπροσώπηση όλων αυτών των διαφορετικών συμφερόντων, αλλά επίση επειδή ακούγονται και διαφορετικέ φωνέ και διαφορετικέ εξειδικευμένε γνώσει που έχουν αυτοί. Και βεβαίω, τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πολύ συχνά εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί μάλλον την εξειδικευμένη γνώση και τι εκθέσει του ILO. Ακριβώ, λοιπόν επειδή πρόκειται για ένα τριμερή οργανισμό, ε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε, ε, θα πρέπει μάλλον να αντιληφθούμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Δεν πρόκειται για έναν οργανισμό, για παράδειγμα, ο οποίο επιβάλλει κυρώσει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τον ΔΟΕ. Η κυρία Τούνιγκα, τώρα εγώ θα έρθω σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Ε, ε, μας ζητήθηκε να εξηγήσουμε πώς συνεργαζόμαστε με τον ΔΟΕ ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πως γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με το ΔΟΕ. Και πιο συγκεκριμένα μας ρωτήσατε τι κάνουμε σε σχέση με την εφαρμογή. Για εκείνους που ίσως να μην το γνωρίζουν, ήδη από το 2017-2018 έγινε μια πολύ ευρία συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία μας και καταλήξαμε μάλιστα σε ένα σχέδιο δράσης με 15 σημεία ε, και κάτι που φάνηκε είναι ότι χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των διεθνών οργανισμών. Και προσπαθήσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την νοοτροπία ε, στη συνεργασία μας με τον ILO για την εφαρμογή των κεφαλαίων GSP στις ε, συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας. Αξιοποίησαμε λοιπόν την τεχνική συνεργασία για όλες τις χώρες που ήδη αναφέρθηκαν, Βιετνάμ, ε, Κυργιστάν και άλλες. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με τον ILO και στο TSD και στο GSP. Για να σας δώσω τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τον τομέα του TSD. Ε, θέτουμε συγκεκριμένο κατάλογο προτεραιοτήτων, δηλαδή θέματα στα οποία θα ήθελε να εστιάσει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το που καταλήγουμε εμείς ως Ένωση στις προτεραιότητές μας, ενημερώνουμε τον ILO. Και βεβαίως γνωρίζουμε ήδη τι συζητήτες στον, ε, στο, στον ILO και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις αλληλοεπικαλύψεις. Αν γνωρίζουμε ότι ο ΔΟΕ πρόκειται να επέμβει σε μια χώρα όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα εργατικής νομοθεσίας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε το, το ίδιο, απλώς ενισχύουμε τις προσπάθειες του ILO. Ε, συνεργαζόμαστε ε, σε αιτήσια βάση με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας δημιουργούνται επίσης και επιτροπές, αξιοποιούμε τη γνώμη ε, τοπικών οργανώσεων ή εξειδικευμένων επαγγελματικών οργανώσεων, τις οποίες προσκαλεί συχνά ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας στις ε, συναντήσεις του. Και επίσης, όπως ήδη ανέφερε και ο συνάδελφος, παρακολουθούμε τις, τα διαμοιβόμενα στις διάφορες επιτροπές του ε, ΔΟΕ και συνεισφέρουμε σε αυτές. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή τη συνεχή και ε, εις βάθος συνεργασία που αξιοποιεί την τεχνική βοήθεια και μετά σε συμφωνίες που περιλαμβάνουν κεφάλαιο GSP έχουμε και συγκεκριμένε ρήτρε για τη δέουσα επιμέλεια. Έχουμε αντίστοιχε για τι περιπτώσει τη Λατινική Αμερική και για την Ασία. Στην περίπτωση τη Λατινική Αμερική έχουμε και συμμετοχή του ΟΑΣΕ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην δεύτερη ε, περίπτωση. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά βοηθάει αυτές τις τρίτες χώρες να υλοποιήσουν τις κατευθυντήριες αρχές για τη δέουσα επιμέλεια. αξιοποιούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τι κατευθυντήριε γραμμέ του ΟΑΣΕ για, του ΟΑΣΑ, για τι πολυεθνικέ επιχειρήσει εδώ. Και είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσα να σας μιλήσουμε πολύ πάθος, γιατί είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία αυτού του σχεδίου δράσης με τα, 17, με τα 15 σημεία που πραγματικά καταφέραμε να υλοποιήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική συνεργασία με τον ΔΟΕ που την είδαμε να εφαρμόζεται στην περίπτωση του Βιετνάμ. Και το είδατε και όταν η Επιστροπή σας επισκέφθηκε τη χώρα, πώς απευθύνονταν οι εκπρόσωποι της χώρας αυτής προς τους εκπροσώπους της, του ILO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας μας ουσιαστικά να τους βοηθήσουμε για την υλοποίηση αυτών των, αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Υπογραμμίζω και εγώ το τελευταίο σημείο που αναφέρατε, Μαδλέν και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Μερικές φορές το κύριο ερώτημα είναι θέμα προσωπικότητων, κατάστασης κάθε χώρας που θεωρούνται ως θεσμοί ουσιαστικά, έχουν παγιωθεί. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Έχουμε και κάποια αρνητικά παραδείγματα φυσικά από την Αμερική που δεν θέλω να αναφέρω, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να σταθεροποιήσουμε, να θεσμοθετήσουμε ή να παγιώσουμε τη συνεργασία ε, εδώ ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά υπό την επιτήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κλείνει αυτή η συζήτηση. Κυρία Κέρτη, θα παραμείνουμε σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. So, next item is the item. Το επόμενο σημείο είναι το 6 Επίσης σημαντικό ζήτημα, πέραν των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έχουμε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία και την επιβολή τους ε, και την παρακολούθησή τους ε, σε τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον περασμένο Δεκέμβριο μια έκθεση για το θέμα αυτό. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση αυτή και να ρίξουμε μια ματιά σε μεγαλύτερο βάθος ε, για την κατάσταση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ε, σε τρίτες χώρες και φυσικά ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η Κίνα ε, τα περισσότερα προβλήματα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορούν την Κίνα φυσικά Οπότε ελπίζω να συζητήσουμε και σε αυτό το πλαίσιο τα προβλήματα που έχουμε προσδιορίσει στην Ινδία, στην Ινδονησία, Ρωσία, Ουκρανία και Τουρκία. Θα δώσω το λόγο στον Πίτερ Κόβατς, τμήματάρχη, που θα μας δώσει μία εικόνα για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω σήμερα την τελευταία έκθεση για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 9 Ιανουαρίου του 2020. Πρόκειται για την τελευταία έκθεση μια σειράς εκθέσεων τις οποίες εμείς εκδίδουμε κάθε δύο χρόνια. Ουσιαστικά επικαιροποιούμε ε, τις ε, εκθέσεις αυτές βάσει της τρέχουσας κατάστασης. Αποτελεί ένα το κομμάτι της ε, προσπάθειας της Επιτροπής για ενίσχυση της προστασίας και της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τον γενικό στόχο πώς συνδέονται η διανοητική ιδιοκτησία στην με την καινοτομία, με την οικονομική ανάπτυξη, με την προστασία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας τώρα συνεργαζόμαστε με την Ευρωπόλ, τις Εθνικές Αρχές Επιβολής ε, και άλλες ε, αρχές και αυτή η συνεργασία δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες και ότι πρέπει να τις περιορίσουμε. Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της έκθεσης που ονομάζουμε την έκθεση των τρίτων χωρών. Είναι να εντοπίσουμε τις τρίτες χώρες όπου η κατάσταση της προστασίας και της επιβολής των δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες. Η ανάλυση αυτή δεν είναι πλήρης όσον αφορά την προστασία και την επιβολή του IPR στον κόσμο η, χώρα με τις προτεραιο... η λίστα με τις προτεραιότητες αναχώρα ε, δεν είναι απόλυτη. Έχουμε συμπεριλάβει στη λίστα αυτή τις χώρες όπου η έλλειψη επιβολής και προστασίας IPR και οι ελλείψεις που υπάρχουν ε, δημιουργούν ε, την μεγαλύτερη βλάβη στα ευρωπαϊκά συμφόραντα. Επίσης, η έκθεση θέλει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους της μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις ε, για τις ε, δυνατότητες που έχουν όσον αφορά τα IPR και τους κινδύνους που διατρέχουν σε ορισμέ, στο πλαίσιο ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες, ωστόσο ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους και τις ε, δράσεις τους για να προστατεύουν τα άειλα αγαθά τους, τα άειλα περιουσιακά τους στοιχεία. Η έκθεση είναι χρήσιμη όπως έχει αποδειχθεί και για αρχές τρίτων χωρών. Ε, ως πηγή πληροφοριών. Η λίστα προτεραιοτήτων ε, χρησιμεύει επίσης και στην Κομισιόν. Μας βοηθάει να εστιαστούμε στους πόρους μας, οικονομικούς και ανθρώπινους, σε ορισμένε χώρες. Έχουμε διάφορες ε, συνεργασίες ή προγράμματα με την Κίνα, την Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική. Μόλι έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συνεργασία στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησία για να υποστηρίξουμε την Αφρική στι προσπάθειε τη να βελτιώσει την κατάσταση αυτή. IPR εκεί. Έχουμε διάφορου διαλόγου με χώρε ε, και εκεί έχουμε συμπεριλαβεί την Κίνα, την Ταϊλάνδη, προσπαθούμε και με την Ινδία και κάποιε άλλε χώρε κατά κύριο λόγο εκείνες που βρίσκονται στη λίστα προτεραιότητας ούτω ώστε να προασπίσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Όσον αφορά τη λίστα προτεραιοτήτων, δεν παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές. Ε, ουσιαστικά η Κίνα έχει παραμείνει ως χώρα νούμερο ένα σε προτεραιότητα. Δεύτερη Ινδία, Ινδονησία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία. Οι χώρες προτεραιότητας τρία είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Σημερινός, η Μαλαισία, η Νιγηρία η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη. Η σειρά κατάταξης και η αιτιολόγηση για την κατάταξη μιας χώρας ε, ως προτεραιότητας 1, 2 ή 3 αιτιολογείται από την κλίμακα και την ε, διαρκή ύπαρξη προβλημάτων στον τομέα της προστασίας και την επιβολή των ε, δικαιωμάτων διανοητικής διεκτησία. Και όπως καταλαβαίνετε η Κίνα είναι αυτή που μας ανησυχεί περισσότερο. Εγώ ήμουν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα. Εκεί κάναμε μια μεγάλη συζήτηση με τους ομολόγους μας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την επιβολή του στην Κίνα και αυτή ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με τα πορίσματα της έκθεσης και αυτό είναι καλό σημάδι για μας. Αυτό σημαίνει ότι ε, πετύχαμε διάνα. Ε, συζητήσαμε ακριβώς τα προβληματικά ζητήματα με, που αφορούν την Κίνα στη χώρα αυτή, ε, στην έκθεση αυτή των τρίτων χωρών και τελικά συμφωνήσαμε ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας και επιβολής στην Κίνα. Πολλά διαφορετικά προβλήματα παρατηρούνται σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον των χωρών προτεραιότητας, ε, επίσης, ε, δημιουργήσαμε και ένα τμήμα για κάποιες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνάψει ή πρόκειται να συνάψει σύντομα ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών και εκεί παρατηρείται ιδιαίτερη ανάγκη παρακολουθήσης της κατάστασης των ΑΠΙΑΡ. Μιλάμε για Καναδά, Νότιο Κορέα, Μεξικό και Βιετνάμ. Επίση, θα παρακολουθεί στενά η Επιτροπή την κατάσταση σε άλλε χώρε όσον αφορά την επιβολή IPR όπου σημειώνονται ανησυχητικά περιστατικά. Δεν είναι στη λίστα προτεραιότητα, αλλά είναι υποψήφιε για να μπουν στη λίστα αυτέ οι χώρε ή ήταν παλιότερα και μόλι έχουν βγει ε, και έχουν μπει σε μια λίστα Προ παρακολούθηση Ισραήλ, Μαρόκο, Παραγουάη, Φιλιππίνες, Νότιο Αφρική, Ελβετία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε σε αυτή την εκθέση είναι ότι εντοπίζουμε χώρες, ε, βασικές τάσεις, βασικά ζητήματα. Οπότε αν κάνετε μια σύγκριση των δύο εκθέσεων, εκείνης που δημοσιεύτηκε πριν από δύο χρόνια με την ε, τελευταία έκθεση, οι χώρες έχουν παραμείνει μέσα σε κρίση ίδιες. Με δύο-τρεις διαφορές. Τα προβλήματα μπορεί να διαφέρουν, ε, διότι καμιά φορά ανακαλύπτουμε νέα προβλήματα και στη τελική ανάλυση έχουμε επιλύσει και πολλά ζητήματα σε χώρε με τι οποίε έχουμε διάλογο και συνεργασία συμπεριλαμβανομένη περίεργω και τη Κίνα. Ε, έχει σημειωθεί πολύ καλή πρόοδο. Παρόλα αυτά, παραμένουν ακόμα προβλήματα. Οι ομολογοί μας αμφισβητούν ε, την παρουσία του στη λίστα Αναρωτιούνται πώς δουλεύουμε, από πού παίρνουμε πληροφορίες και φυσικά τι τους λέμε εμείς ότι τα γεγονότα και τα στατιστικά στοιχεία σπάνια ψευδόνται και ότι η εργασία μας βασίζεται κυρίως σε δημόσια διαβούλευση ότι όλοι, ε, δηλαδή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δικαιούχοι δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, οποιοδήποτε άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί προστασίας των καταναλωτών, όλοι μπορούν να συμβάλλουν και να στείλουν πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η δουλειά μας, η οποία επίσης βασίζεται και σε διάφορες μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΕΟΕΠΗ συμβάλλει πολύ ε, μελέτες του ΩΣΑ, συνεργαζόμαστε και με πολλούς άλλους οργανισμούς. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο και εκεί σε θέματα παραποιημένων αγαθών τα γεγονότα είναι καθαρότατα και οι τάσει επίσης. Έχουμε δηλαδή μία στιβαρή βάση και για την έκθεση και για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, σίγουρα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να προσπαθούμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό είναι ο βασικό στόχο τη εκθέση αυτή, Να σημειωθεί η πρόοδο και να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτές τις Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεργασία μας μαζί του, στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασία μα, στο πλαίσιο των διαλόγων μα, των ομάδων εργασία και διαφόρων άλλων ε, τρόπων συνεργασίας που έχουμε δημιουργήσει ή που θέλουμε να δημιουργήσουμε με τις προβληματικές χώρες θα θυμάστε ότι είχαμε και μια άλλη σημαντική έκθεση που ήταν ο κατάλογος παρακολούθησης για παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα που δημοσιεύουμε κάθε δύο χρόνια. Η τελευταία τέτοια έκθεση δημοσιεύτηκε πέρυσι δηλαδή και θέλουμε να δημοσιεύσουμε, να δημοσιεύσουμε την επόμενη στα τέλη του 2020. Πρόκειται για μια λίστα πλατφόρμων αγορών ουσιαστικά, εταιριών και αγορών στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου που υποψιαζόμαστε ότι εμπλέκονται με θέμ, προβλήματα παραβίασης ε, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι της εκθεσής μας και θα ξεκινήσουμε σύντομα την δημόσια διαβούλευση για την έκθεση αυτή. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της εργασίας μας. Θα συνεχίσουμε να σας διατηρούμε ενήμερους λοιπόν για τις προσπάθειές μας και φυσικά θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσά πώ θεωρείτε θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την εργασία μα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Μπορσουά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την λεπτομεριακή έκθεση και εισήγηση. Όταν μιλάμε για αυτές τις αξιολογήσεις και τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούω ότι η Κίνα είναι το πρωταρχικό τους μέλημα. Έγιναν ε, επισκέψεις στην Κίνα και συμφωνήθηκε να υπάρξει καλύτερη προστασία. Το ερώτημά μου είναι ποια συγκεκριμένα μέτρα και συμφωνίες έχουν επιτευχθεί και κάτι άλλο. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες όταν μιλάμε για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Θεωρείτε ότι βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαμε να έχουμε αμεσότερη προστασία σε χώρες ανά τον κόσμο. Και επίσης η Επιτροπή έχει ε, μία υπηρεσία εφαρμογής του πλαισίου αυτού. Θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και την διανοητική ιδιοκτησία μέσω αυτού του μηχανισμού. Ως προς το Βιετνάμ, το οποίο επισκέφθηκα όλας, είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, έχουν ε, οργανωθεί προγράμματα, βέλτιστες πρακτικές, ανταλλαγές επ' αυτών και ούτω καθεξής, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Άρα η Επιτροπή είδε έμπρακτα αποτελέσματα Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την έκθεση αυτή και την εισήγηση. Θα ήθελα να υποβάλω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στην έκθεσή σας μιλάτε για τη σημασία των ε, τελωνιακών αρχών μέσα στα πλαίσια του ελέγχου και πολλές ε, χώρες δεν έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ως προς το κυρωτικό πλαίσιο, τις κυρώσεις δηλαδή που επιβάλλονται, ε, δυστυχώς ε, είναι πολύ, ε, είναι ελαχιστότερες κατά πολύ της βλάβης που προκαλείται από τις παραχαράξεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, δεν υπάρχει μία τελωνιακή αρχή, ενιαία τελωνιακή αρχή και δεν υπάρχει ένας κυρωτικός μηχανισμός ο οποίος να μπορεί να εφαρμοστεί σφαιρικά. Τι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσε να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, και θα τελειώσω με αυτό, μιλάμε για τη ε, ε, σημασία των ενδείξεων και υποδείξεων που έχουμε για να καταπολεμήσουμε τις ε, παραχαράξεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει μία έκθεση σε σχέση με το γεωγραφικό προσδιορισμό και τις ε, μικρές βιοτεχνίες καθώς και τις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παραχάραξη ιδιαίτερα όταν προέρχεται από την Κίνα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ολιστικά αυτό το θέμα των παραχαράξεων. Έχετε κάτι να μας υποδείξετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιωρή. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να πω ότι με, με εξέπληξε το γεγονός ότι η Ουκρανία βρίσκεται στις προτεραιότητες υπαριθμών 2, γιατί από όσο ξέρω είναι η μόνη χώρα που είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος και έχουμε και μια συμφωνία σύνδεσης. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι τα ευρήματα της Επιτροπής σε σχέση με την Ουκρανία. Κατά πόσο οι Ουκρανικές αρχές θέλουν να συνεργαστούν επί του θέματος, έχει αλλάξει η νομοθεσία ή θα έχουμε θετικά βήματα ως προς την ε, εφαρμογή αυτού του πλαισίου, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και πώς εφαρμόζεται το όλο πλαίσιο στην Ουκρανία. Η κυρία Καβατσίνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Γνωρίζετε ε, ποια είναι τα δεδομένα σε σχέση με την Αντισαμπέμπα, σε σχέση και με τους ε, αναπτυξιακούς στόχους Υπάρχει και το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τη διάδοση της τεχνολογίας στις υποανάπτυξη χώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς η Επιτροπή θα εφαρμόσει αυτή την ατζέντα της Μπέμπα έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και το περιβάλλον αλλά και τη διανοητική ιδιοκτησία καθώς και θέματα ε, υγείας. Ξέρετε ότι τα γενώσιμα πολλές φορές σώζουν ε, ζωές και αυτό αφορά και περιβαλλοντικά αγαθά, διότι ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτά τα θέματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών. Ε, η συνάδελφος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση μας είπε και ο Πρόεδρος ότι αυτό το θέμα είναι ύψης της σημασίας για την οικονομία μας και εσείς ε, ακριβώς ε, το ίδιο είπατε. Ε, αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών. σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μπουρζουά, συμφωνώ ότι δηλαδή μας ενδιαφέρει η εφαρμογή του πλαισίου σε σχέση με την αρχή επιθεώρησης. Η Επιτροπή ε, θα πρέπει να μας πει κατά πόσο υπάρχουν ανταλλαγές και όπως και η κυρία Ροντρίγκε, θα ήθελα ε, να μας πείτε ποιες είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις, όχι βεβαίως στον αγροτικό τομέα και ως προς τις ΜΜΕ θα τις βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισήγηση αυτή. Υπάρχει και το παράδειγμα της Ουκρανίας, διαβάζοντας την έκθεσή σας. Επειδή δεν κατανοούμε πώς έχει η νομοθεσία σε αυτή τη χώρα και πού προς τα που κινούμαστε, δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να συναυθεί μια συμφωνία σε σχέση με την αντιμετώπιση των ε, παραχαράξεων. Δηλαδή, πώς έχουν οι διαβουλεύσεις για να υπάρχει εφαρμογή μηχανισμών προστασίας της ε, διανοητικής ιδιοκτησίας. Ποιες είναι οι υποδείξεις σας για να έχουμε πιο αξιόπιστες ε, μετρήσεις στην οικονομική συνεργασία με τις τρίτες χώρες που θα πρέπει να ενταχθεί στην Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Αυτό αφορά και τη Βραζιλία και την Αργεντινή σε σχέση με τις προτεραιότητες υπαριθμών 3. Ποιες είναι έμπρακτα οι προτάσεις σας. Δεύτερον, σε σχέση με την Κίνα, η Κίνα ενέκρινε μία νομοθεσία η οποία ε, στην ουσία συγχαίει το πλαίσιο της παραχάραξης με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στον τομέα των εξαγωγών και την νέα εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Και το Βιετνάμ το αναφέρεται επικριτικά κατά κάποιο τρόπο. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα εν ώψη των συμφωνιών. Γιατί διαφορετικά πάλι θα σκοντάψουμε στο ίδιο θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ουσιώδης προστασία ως, με, ως προς τις παραγωγικές διαδικασίες αντιμετώπισης των μελλοντικών προκλήσεων στα πλαίσια της ψηφιοποίησης. Ο κύριος Ντάντη. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά καθυστέρησε η πτήση μου, γι' αυτό ήρθα και αργά. Αυτό είναι θέμα στρατηγικής ε, σημασίας που προανέφεραν και ορισμένοι συνάδελφοι, συνάδελφοι ως προς τους, τις γεωγραφικές ενδείξεις ε, που δεν άπτονται του τομέα της διατροφής. Μιλάμε για μη γεωργικά προϊόντα τα οποία ε, εποπτεύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει η Επιτροπή να προβάλλει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, διότι είχαμε 600, 653 ψήφους υπέρ και περίπου 50 κατά, 50 κατά και 50 αποχές και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι τα προσκόμματα που θέτουν ορισμένες χώρες για να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία και τις βιοτεχνίες ιδιαίτερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στεναρά την Κίνα, διότι μέσω τελωνιακών αρχών στην προηγούμενη θητεία σε μια αποστολή στην Κίνα είδα ότι έχουμε ένα ουσιώδες πρόβλημα όχι ως προς την νομική προστασία από πλευράς ε, Κίνας της διανοητικής ιδιοκτησίας. Αλλά πολλές επιχειρήσεις μας λένε ότι υπάρχουν αποφάσεις κινέζικων δικαστηρίων σε σχέση με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που αγνοούνται από τις κινέζικες αρχές. Δηλαδή τα διπλώματα έβρεση τεχνίας πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται, δεν υπάρχει έλεγχος και δεν υπάρχει έλεγχος και εποπτεία. Αυτό αφορά και την παραχάραξη και την πνευματική ιδιοκτησία γενικότερα. Διαφορετικά ακυρώνουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος με συγκεκριμένες απαντήσεις από τις ε, κοινωνικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά είναι τα στοιχεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω, θέματα προς αντιμετώπιση. Ευχαριστούμε πολύ. Ερώτηση και από εμένα, σύντομη, σε σχέση με κάτι που αναφέρεται στη σελίδα 14. Τρεις ερωτήσεις μάλλον. Πρώτον, Υποβάλλετε κάποιες εκθέσεις στα μέλη, λέτε, του Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου, του ΠΟΕ. Ιδιαίτερα εκείνε τι χώρε, λέτε, στι οποίε συμπίπτουν οι θέσει μα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι αντιδράσει αυτών των χωρών, ιδιαίτερα σε σχέση με τι ε, παρεμβάσει μα για χώρε όπω η Κίνα ή άλλε. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι εάν υιοθετηθούν επιπλέον κανόνες για τη διανοητική ιδιοκτησία, στο, στους κανόνες του ΠΟΕ, στο rulebook του ΠΟΕ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες συγκρούσεις με ορισμένα κράτη-μέλη του ΠΟΕ. Δηλαδή να προσπαθήσουν να το σταματήσουν. Τρίτον, αναφερθήκατε στην ε, διαμάχη στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την Κίνα και Κατά πόσον θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να ενισχύσουμε την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Το όργανο προσφυγών του ΠΟΕΝ. Στο συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που άργησα, χρειάστηκε να συναντηθώ με εκπρόσωπο ε, της γερμανικής κυβέρνησης, αλλά για πολύ διαφορετικό θέμα. Ε, εγώ θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα σε σχέση με το πρώτο κεφάλαιο της Συμφωνίας Ευρω... ε, συγγνώμη, ε, Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αναφέρεται στη διανοητική διοκτησία. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται μετά στην μεταφορά τεχνογνωσίας. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτή τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή και Κίνας όσον αφορά την εφαρμογή της και την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ε, και επίσης θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στα δικά μας πρότυπα ή ταιριάζει περισσότερο στις πολιτικές επιδιώξεις του Πρόεδρου Τραμπ. Το δεύτερο μου ερώτημα έχει σχέση με τις προστατευμένες γεωγραφικές ονομασίες. Εδώ αναφέρεται ότι η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντικό αίτημα από άλλον εμπορικό εντέρο για την αναγνώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης δεν θα υπονομεύσει τις δυνατότητες ε, των ε, επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες στη χώρα αυτή. Πρόκειται για το άρθρο 1.15 ε, από τη Συμφωνία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή: Πώ αυτή η συμφωνία τη Κίνα με τι ΗΠΑ θα επηρεάσει την πιθανή συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα. Σα ευχαριστούμε να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερως που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το έργο μας και ιδιαίτερα για το ζήτημα της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Επιτροπή σας. Δεν με εκπλήσει η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε όσο καλύτερα μπορώ. Ας ξεκινήσουμε με την Κίνα που είναι και το πιο εύκολο. Λοιπόν, παραμένει η χώρα πρώτης προτεραιότητας, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Έχουμε την εξή προσέγγιση. Βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μας δίνουν τα ενδιαφερομένα μέρη και από αυτές έχουμε καταπτύσσει τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτον, την νομοθεσία. Δεύτερον, η ε, καταχωρήση εμπορικών σημάτων με κακή τυπίστη. Ορισμένοι ομιλητέ αναφέρθηκαν σε αυτό. Αρχικά είχαμε εστιαστεί στο, στα trademarks, ε, ε, στα εμπορικά σήματα, αλλά τώρα πλέον μιλούμε και για άλλο είδες, ε, άλλα εργαλεία πρωτοστασία της διανοητικής ιδιοκτησία, όπως οι πατέντες ή τα, τα, τα υποδείγματα, utility models. Τρίτον είναι το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας, γιατί ξέρουμε ότι αν η νομοθεσία μένει στα χαρτιά δεν προσφέρει τίποτα. Και τέταρτον, εξίσου σημαντικό, ε, είναι η εξαναγκαστικές μεταφορές τεχνογνωσίας. Ένα πρόβλημα το οποίο ε, έχουμε επισημάνει και με το οποίο έχουμε συγκρουστεί με τις αρχές της Κίνας ε, εδώ και πολύ καιρό και στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Στον τομέα της νομοθεσίας έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την πλευρά της Κίνας. Υιοθέτησαν διάφορους νόμους, για παράδειγμα άλλαξαν την νομοθεσία του σε σχέση με τα εμπορικά μυστικά, άλλαξαν την νομοθεσία του σε σχέση με τα εμπορικά σήματα, τώρα η διατύπωση, η νέα της νομοθεσίας είναι ικανοποιητική. Συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα με την νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις πατέντες. Και αυτό βεβαίω δημιουργεί προβλήματα σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει οι οποίε προσπαθούν να ε, υπερασπιστούν κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνία που διαθέτουν στην Κίνα. Και βεβαίω οι εταίροι μα με του οποίου συνομιλούμε από την Κίνα δεν έχουν μπορέσει ακόμα να μα ενημερώσουν πότε σκοπεύει η χώρα αυτή να υιοθετήσει μια νέα νομοθεσία για το ε, δίκαιο ευρεσιτεχνία, για το copyright. τουλάχιστον για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία γνωρίζουμε ότι μέχρι το τέλο του 2020 θα υπάρξει πρόεδρο. Για το copyright δεν έχουμε κάποια αντίστοιχη πληροφόρηση. Τώρα για τι εγγραφέ κακή την πίστη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την προστασία των εμπορικών σημάτων και των διακριτικών τίτλων Μιλώντας με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Σανγκάη την προηγούμενη εβδομάδα, όλες μου επιβεβαίωσαν ότι μπορεί να έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων για τη διανοητική ιδιοκτησία σε μεγάλες πόλεις όπως το Πεκίνο, η Σανγκάη. Ε, ε βελτιώθηκαν τα πράγματα, μεν, αλλά οι αποφάσεις που εκδίδουν τα περιφερειακά δικαστήρια διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και, είναι, και υπολείπονται πολύ των προτύπων. Είναι σε πολλές περιπτώσεις κακής ποιότητας αυτές οι δικαστικές αποφάσεις από τα περιφερειακά δικαστήρια. Τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Οι επικρίσεις που ασκούμε στην έκθεσή μας εστιάζονται στα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου και εστιάζονται δηλαδή στις τρίτες χώρες κυρίως, ιδιαίτερα σε σχέση με την Κίνα. Διαπιστώνουμε ότι έχουν αυξηθεί οι ποινές που επιβάλλει η χώρα αυτή όταν υπάρχει παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησία σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα όταν υπάρχει παραβίαση εμπορικού σήματος. Και το επίπεδο αυτών των κυρώσεων που πλέον επιβάλλει η Κίνα έχει αρχίσει να ικανοποιεί και τους δικούς μας ε, ενδιαφερόμενους. Όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, στον τομέα των εμπορικών μυστικών έχουν υπάρξει νέες ρυθμίσεις. Έχουμε λοιπόν και νέα νομοθεσία σε σχέση με τα εμπορικά σήματα στο πλαίσιο αλλαγών που έγιναν στην νομοθεσία για τον ανταγωνισμό. Πρέπει να δούμε όμως πώς αυτές οι αλλαγές στην νομοθεσία εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Κίνα, στην αχανή έκταση της Κίνας. γνωρίζουμε βέβαια ότι το οικονομικό κέντρο της χώρας αυτής ε, εστιάζεται κυρίως στην Ανατολή. Αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι σημαντική σε ολόκληρη τη χώρα. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε γενικέ γραμμέ η πρόοδο που βλέπουμε στην Κίνα έχει σημειωθεί ακριβώ επειδή η Κίνα αντιλήφθη ότι αυτό είναι και προς δικό τη όφελο. Έχει αρχίσει να γίνεται πλέον μια υπερδύναμη στον χώρο τη διανοητική ιδιοκτησία. Υπάρχουν πλέον πολλέ κινοζικές επιχειρήσει οι οποίε ε, γράφουν ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και, και αποκτούν δικαιώματα ε, διανοητική ε, ιδιοκτησία. Πρόκειται μια, μια χώρα η οποία επενδύει πολλά στην έρευνα, προσπαθεί να γίνει υπερδύναμη στον τομέα αυτό. Και άρα έχει καταλάβει ότι είναι προ το συμφέρον τη να βελτιωθεί. Όμω συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των ξένων επιχειρήσεων στην Κίνα σε σχέση με τι κινέζικε. Αυτό παραμένει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ασκώντα πίεση. Και τώρα, η πρώτη αξιολόγηση που κάνουμε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα θα λέγαμε ότι είναι θετική. Γιατί πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση, ασκεί μια πίεση προ την Κίνα να εφαρμόσει την νομοθεσία τη για την προστασία τη διανοητική ιδιοκτησία με τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσει, που δεν θα ε, ε, ασκεί διακριτική μεταχείριση εναντίον των ξένων επιχειρήσεων. Ε, υπ' αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίω, Μόλις στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας δημοσιοποιήθηκε το κείμενο της συμφωνίας, άρα συνεχίζουμε να κάνουμε την ενδική μας αξιολόγηση. Αλλά μια πρώτη αντίδραση από τη δικιά μου πλευρά θα έλεγα ότι είναι θετική, γιατί ε, είναι μια συμφωνία που ασκεί πίεση στην Κίνα να βελτιωθεί στον τομέα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. Βεβαίως, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό είναι ότι γεγονό ότι ε, ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσει με την Κίνα για τη Συμφωνία για την Προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων, GI. Τώρα, θεωρούμε ότι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων έχει ολοκληρωθεί. Άρα δεν θεωρούμε ότι η άλλη συμφωνία που έκαναν με τι ΗΠΑ μα επηρεάζει σε οποιοδήποτε βαθμό. Αυτή είναι βέβαια η δική μας αξιολόγηση των πραγμάτων. Θα δούμε κατά πόσον θα επιβεβαιωθεί. Αλλά πάντως οι διατάξεις στη δική μας συμφωνία είναι ξεκάθαρες. Και γυρίζω στον παρόδο αυτό που πάντα προσπαθούμε να εξηγούμε στους εταίρους μας είναι ότι η επιδίωξή μας δεν είναι να δημιουργούμε προσκόμματα στο εμπόριο ή προσκόμματα στις εξαγωγές άλλων χωρών. Αυτό που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε με τις ε, διατάξεις για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις είναι να προστατεύουμε τα ονόματα, να προστατεύουμε τις γεωγραφικά προστατευόμενες ονομασίες αγροτικών και άλλων προϊόντων. Ε, αυτό είναι κάτι βασικό στην ευρωπαϊκή μας νομοθεσία και φυσικά η Επιτροπή θα συνεχίσει να την προστατεύει στη σχέση της με τις τρίτες χώρες. Τώρα, Εάν υπάρχουν κάποιες γρήγορες λύσεις, με ρωτάτε, εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό στους τομείς ε, που συζητούμε. Οι διαδικασίες συνήθως είναι μακροχρόνιες και έτσι μακροχρόνιες έχουν υπάρξει και οι συζητήσεις μας με την Κίνα. Θα έλεγα το Μάρτιο, αν δεν απατώμε, έχουμε τη 15η επέτειο της λειτουργίας ε, της Επιτροπής Δομημένου Διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ενώ υπήρχαν και άλλα προγράμματα που είχαν ξεκινήσει ακόμα παλαιότερα. Ε, μετά λοιπόν από αυτά τα 15 χρόνια μπορούμε πια να πούμε ότι έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος, χωρίς αυτό να είναι αναγκαστικά εντυπωσιακό, αλλά ε, τουλάχιστον μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ε, σημειώθηκε πρόοδος και τα πράγματα βελτιώθηκαν. Τώρα, σε σχέση με το Βιετνάμ. Η Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου συμπεριλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για τη διανοητική διοκτησία με ουσιαστικές διατάξεις Βεβαίω θα τεθεί και πάλι το θέμα τη ουσιαστική εφαρμογή και από την πλευρά μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει να παρακολουθήσει την εφαρμογή τη συμφωνία. Πέραν από τη συμφωνία, ε, σα το ανέφερα και προηγουμένω, έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συνεργασίας ε, με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασία συνολικά για την προστασία τη διανοητικής ιδιοκτησία. Το βασικό στόχο αυτού του προγράμματο συνεργασία το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η UIPO, είναι λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες αυτής της περιοχής να εφαρμόσουν τις συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει μαζί τους. Κάνουμε ό,τι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε με τις χώρες αυτές, πιστεύω, και από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με τη Βιετνάμ θα την παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενά έτσι ώστε να εφαρμοστεί. Τώρα, γεωγραφικές ενδείξεις μη αγροτικών προϊόντων. Το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, δεν αφορά την DigiTrade, είναι ο Επίτροπος Μπρετών αρμόδιος ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις που δεν είναι γεωργικές. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι συμμετέχουμε ήδη, ακόμα μάλλον στις εργασίες, ε, γίνονται διερευνητικές εργασίες. Εξετάζονται βασικά ζητήματα για την εισαγωγή των μη γεωργικών ε, γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για μας, για την DigiTrade και για τους διαπραγματευτές, βασικό στοιχείο είναι ότι θα μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα να συμπεριλάβουμε μη γεωργικές ε, γεωγραφικές ενδείξεις, διότι πολλοί μας εμπορικοί εταίροι έχουν τέτοιες μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις. Θα δημιουργούσε μια καλύτερα βάση για να διαπραγματευτούμε με αυτές τις χώρες και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις που θέλουμε να προστατεύσουμε θα προστατευτούν σωστά εφόσον δώσουμε κάποιο σωστό αντάλλαγμα. Και αυτό θα μας βοηθούσε πολύ στις διαπραγματεύσεις μας. Αλλά φυσικά Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ πιο μεγάλα και σημαντικά θέματα. Ωστόσο, η Νέα Επιτροπή εξετάζει ένεργα το ζήτημα αυτό της εισαγωγής των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων. Για την Ουκρανία. Γιατί είναι η Ουκρανία στον κατάλογο ως μία από τις κύριες χώρες, διότι εξακολουθούμε να έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα στην Ουκρανία όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ακόμη και την ε, εισαγωγή τους. Η Ουκρανία επί της αρχής ευθυγραμμίζεται απόλυτα βάσει υποχρεώσεών της, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Σύνδεσης. από αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί στη συμφωνία έχει εφαρμόσει ωστόσο ελάχιστα η Ουκρανία. Πραγματοποιείται τακτικά συζητήσεις με τις Ουκρανικές αρχές και γίνεται μια προσπάθεια να ασκήσουμε πίεση, αλλά η διαδικασία λήψη αποφασών χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντικά προβλήματα. Δεν περνούν νόμοι ε, από το Κοινοβούλιο και εκείνοι που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο τελικά δεν υλοποιούνται και σωστά. Εμείς στην έκθεση αναφέρουμε σαφώς ε, ότι εκφράζονται δυστυχώς πολύ σημαντικές ανησυχίες για την Ουκρανία. Συνεχίζουμε βέβαια να συνεργαζόμαστε μαζί τους και να τους υποστηρίζουμε ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε θέματα επιβολής των δικαιωματών διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε ούτε καν να τους πείσουμε ε, να τους πάμε στις ε, χώρες ε, προτεραιότητας 3 φέτος, διότι παρατηρείται απόλυτη έλλειψη προόδου. Πάμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια θέματα, κάθε χρόνο βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο. Πώς θα διασφαλίσουμε τώρα ότι θα σημειώσουν κάποια πρόοδο. Είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Εμεί φυσικά κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί όσον αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να επιμένουμε, να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε βοήθεια. Τώρα δυστυχώς, μάλλον αποτελεί γεγονό ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις ε, στη θέση τους, ούτε να τους επιβάλλουμε αποφάσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ε, η κυβερνητική αρχή που ευθύνεται για τη διανοητική διοκτησία κάνει προσπάθειες, έχει καλή θέληση, αλλά πολύ συχνά απλά δεν περνάνε οι νόμοι ή αν εγκριθούν τελικά κάποιοι νόμοι που συνέβη με μία από τις πρόσφατες νομοθεσίες που αφορούσαν το copyright ξαφνικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές αντίθετες προς το πνεύμα της δικής μας συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία. Οπότε ναι, η Ουκρανία παραμένει ένας ε, μεγάλος πονοκέφαλος για μας σε θέματα επιβολή δικαιωμάτων πνευματική διεκτησία. Η μεταφορά τεχνολογία σε αναπτυσσόμενε χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριζε ανέκαθεν τη μεταφορά τεχνολογία σε αναπτυσσόμενε χώρε. Την ενθαρρύνουμε ενεργά. Επίση, εργαζόμαστε στο πλαίσιο του σχετικού, της Σχετικής Επιτροπής ε, στον ΠΟΕ, όπου γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για την μεταφορά τεχνολογίας. Υποστηρίζουμε δηλαδή το θέμα επί την αρχή, αλλά όχι την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας σε ορισμένε χώρες ή την, ε, αυτοί που μπορούν να επιβάλλουν ορισμένες ε, χώρες σε ορισμένε επιχειρήσεις. Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, ε, ένα σημαντικό στοιχείο, διότι πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικά, μια εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επενδύσει και θεωρεί ότι τα δικαιώματα της, ε, ε στη διανοητική διεκτησία θα είναι ασφαλή ακόμα και αν μεταφέρει τεχνολογία, θα πάνε σε εκείνη τη χώρα και θα δραστηριοποιηθούν εκεί. Τι προσπαθούμε εμείς αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της ε, νέας δράσης ε, ε, στην Αφρική για τα πνευματικά δικαιώματα, για τα δυνατικά δικαιώματα, είναι να ενισχύσουμε τις προθέσεις αυτές των αφρικανικών χωρών να επιβάλλουν, να εφαρμόσουν τα δικαιώματα δυνατική ιδιοκτησίας. Η δραστηριότητα αυτή δεν νομιάζει με αυτήν που χρησιμοποιούμε στην Κίνα, για παράδειγμα. Διότι στην Κίνα το πρόβλημά μας βασίζεται στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και ασκούμε πίεση στους κλάδους όπου έχουμε συμφέροντα ως Ευρώπη και θέλουμε να αλλάξουν τους νόμους, ε, τη στάση τους και τις πρακτικές τους οι Κινέζοι. Στην Αφρική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά διαφορετική δυναμική. Εκεί θέλουμε να συνεργαστούν ενεργά μαζί μας, ούτω ώστε να προσδιορίσουμε από κοινού τις ανάγκες τους. Και επίσης μπορεί να γνωρίζετε ότι στην, ε, σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ε, αποτελούν σημαντικό πυλώνα. Έχει αναγνωριστεί και από τους ίδιους ε, και έχουν ήδη αρχίσει οι αφρικανικέ χώρε να συζητούν και να διαπραγματεύονται το πρωτόκολλο δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία για μια ολόκληρη παν-αφρικανική ε, εμπορική περιφέρεια. Και εμεί του παρέχουμε υποστήριξη σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν του επιβάλλουμε τίποτα, επαναλαμβάνω. Είμαστε στη διάθεσή του για να του βοηθήσουμε στου τομεί εκείνου όπου αισθάνονται ότι υπάρχει ανάγκη. Και φυσικά πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τι δικέ μα ε, ε, με τους δικούς μας ε, ε, χρήσεις και με τα δικά μας συμφέροντα. Αλλά όπως είπα, την αποφάση τη λαμβάνουν οι αφρικανικές χώρες τελικά. Τι θα κάνουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάντα ένα σημαντικό θέμα, διότι οι μεγάλες εταιρείες μέσα στι άκρε ξέρουν πώς να προστατεύσουν τα δικαιώματα δυνατικής ιδιοκτησία τους. Έχουν τους οικονομικούς πόρους και τους ανθρωπίνους πόρους για να μπορέσουν να κυνηγήσουν κάποιον δικαστικά, να προστατεύσουν τα άειλα τους περιουσιακά στοιχεία. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις όχι. Και έτσι έχουμε ξαφνικά, έχουμε δημιουργήσει διάφορα help desk σε διάφορε χώρε ε, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, σε χώρε όπω την Κίνα, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ιαπωνία όπου δεν υπάρχει θέμα προβλημα, ε, δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Προσπαθούμε μαζί με την DigiGrow να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα ε, γραφείων βοήθειας για τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αυτά τα γραφεία βοηθούν να παρέχουν γνώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, πληροφορίες, μερικέ φορέ και βασικές που δεν γνωρίζουν για τις χώρες, για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα διανοητική τους ιδιοκτησία εκεί και άλλα ζητήματα. Για τον ΠΟΕ, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Όπω είπατε πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, συζητάμε με χώρε παρόμοια νοοτροπία, διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία. ειδικότερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου αλλά ο οποίο παραμένει αργός οργανισμό, Εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ χωρών ομοιάζουσα νοοτροπία και αναπτυσσόμενων χωρών όπω η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιο Αφρική, η Κίνα και κάποιε άλλε. Εγώ θα συμπεριλάμβανα και τη Ρωσία σε αυτές. Είναι δύσκολη λοιπόν η συζήτηση. Τώρα, τι προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε σε αυτό το συμβουλευτήριο του ΠΟΕ, να συνεργαστούμε σε κάποια ζητήματα πολύ συγκεκριμένα που ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε κάποια μικρή πρόοδο. Αφορούν κυρίως τις βέλτιστες πρακτικές, την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών Όσον αφορά δηλαδή τις νομοθετικές εξελίξεις, φοβάμαι ότι στην παρούσα χρονική στιγμή είναι ελάχιστε οι δυνατότητες που έχουμε να καταλήξουμε σε νέους ε, νομικά δεσμευτικούς κανόνες στον ΠΟΕ. Η μόνη εξαίρεση όπου ελπίζουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ να έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες είναι, αφορά αυτό τις πρωτοβουλίες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με κάποιες άλλες χώρες με την Ιαπωνία και ακόμα και με τη ΣΥΠΑ προσπαθώντας να επιλύσουμε κάποια ζητήματα όπως την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας αλλά και κάποια άλλα ζητήματα που κατά την άποψή μας είναι αναγκαία για να συνεχίσει ο τις εργασίες του. Όπως είπατε, ναι, δεν υπάρχει δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, όργανο προσφυγών. Όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για την επαναλειτουργία αυτού του οργάνου και μια εναλλακτική λύση επίσης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι ότου το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο να αποκατασταθεί. Ελπίζω λοιπόν να σημειωθεί κάποια πρόοδος στο άμεσο μέλλον για τα ζητήματα αυτά. Ελπίζω να απάντησα μέσα σε άκρες της ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thanks Σας ευχαριστώ πολύ. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Άρα τελειώνουμε και με το θέμα υπαριθμών 6 που ήταν άκρος ενδιαφέρον. Και τώρα έχουμε την κατάσταση προόδου των ενεξελίξη τριμερών διαπραγματεύσεων. Έχουμε μία τέτοια διαπραγμάτευση μακροχρόνια. Είναι ο κανονισμός διτής χρήσης της 13 Νοεμβρίου, στον τελευταίο τριμερί, υπό τη φιλανδική Προεδρία δεν επιτελέστη πρόοδος καταληκτικής υφής. Και τίποτα δεν επετεύχθη. Και η κατάσταση είναι τραγική, συνάδελφοι. Υπάρχει η, τεχνολογία εποπτείας ε, προς τρίτες χώρες που εξάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα μέλη της. Ε, κατά τα τέλη Δεκεμβρίου μπορέσαμε να ελέγξουμε το πρόγραμμα ε, εποπτείας της Τουρκίας που χρησιμοποιείται στην Τουρκία και βασίστηκε σε λογισμικό από τη Γερμανία με μικροαλλαγές και παρήχθη το 2016. Πρόκειται λοιπόν για ένα σχετικά νέο λογισμικό. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί το Συμβούλιο αποφεύγει τη συζήτηση ενδεχομένων λύσεων. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν έχω ιδέα για το τι θα κάνει το Συμβούλιο στο εγγύς μέλλον. Θα το συζητήσω αυτό το θέμα αύριο το πρωί με τον Κροάτι Υπουργό Εμπορίου, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο μετά από πέντε χρόνια, ίσως και έξι. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Ο κύριος Μπούχνερ, ο εισηγητής, είναι παρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Νομίζω ότι είπατε τα πιο σημαντικά στοιχεία, σε αυτά αναφερθήκατε. Θα ήθελα να πω ότι πρόσφατα μία φλαμανδική εταιρεία ε, πούλησε, πούλησε ένα λογισμικό στην Κίνα, ε, ένα σύστημα αναγνώρισης και μας είπαν ότι δεν απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την επίγουσα ανάγκη επίλυσης του ζητήματος. Θα μπορούσα να συνεχίσω εσαΐ e με άλλες υποθέσεις όπου χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή τεχνολογία σε χώρες όπου παραφιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμάμαι έναν προσωπικό μου φίλο στο Ιράν θυμάμαι και ε, τα βασανιστήρια, τις ε, σεξουαλικές οχλήσεις και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και το, την έκθεση του Human Rights Watch του 2020 που αναφέρεται στο ε, Brexit και επειδή ακριβώς υπάρχει διχογνωμία ως προς το μεταναστευτικό καθώς και άλλα ζητήματα είναι δύσκολο να φτάσει σε μία κοινή θέση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία παρά το γεγονός ότι στην αλληρία Σουδάν, ε, ε, ε, Λίβανο, Βολιβία, Ρωσία και Χονγκ Κονγκ οι άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους για να δια, δια μαρτυρηθούν. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η πολύ περιορισμένη υποστήριξη από τις κυβερνήσεις και είναι λυπηρό για το Συμβούλιο και για την Ευρώπη. Ελπίζουμε να βελτιωθεί η κατάσταση με τη νέα Προεδρία. Ευχαριστούμε πολύ. Σχόλια. Ο Μία ερώτηση. Τι θα κάνει η Επιτροπή μας σε σχέση με την εξέβρεση μιας λύσης. Εμείς ε, τι follow-up προτείνουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε ε, δυνατότητες ε, επιβολής κυρώσεων κατά του Συμβουλίου. Θα το συζητήσουμε αύριο με, τη, με τον εκπρόσωπο της νέας Προεδρίας και διαφορετικά θα πρέπει να συνταχθεί ε, μια άλλη πρόταση ψηφίσματος, ένα άλλο ψήφισμα και να ε, διαβιβαστεί στο Συμβούλιο. Μα λίγες είναι οι χώρες που αντιτάσσονται σε αυτή τη συμφωνία. Νομίζω θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε αυτές τις χώρες. έτσι ώστε να μην αντιστέκονται και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε την ε, μέγιστη ε, δυνατή πλειοψηφία στο Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς ε, έχουμε την τροχοπέδη της ομοφωνίας. Χέλμουτ, ρώτησα γιατί στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχουμε το ίδιο θέμα σε σχέση με το δικαίωμα σύστασης ερευνητικής επιτροπής. Επιτροπών έρευνας δηλαδή στο Κοινοβούλιο, δηλαδή και με ε, ειδική, σε, με περίπτωση ειδική πλειοψηφίας θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μία λύση. Ίσως θα πρέπει το όλο θέμα να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε την Κροατική Προεδρία και αυτός είναι ο μόνος δρόμος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά. Εντάξει, θα το αναφέρω. Ωραία. Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν στις 5.30. Ακόμα είναι 5. Μπορούμε να ζητήσουμε τη, από τις πολιτικές ομάδες να μας πούν κατά πόσο μπορούμε να αρχίσουμε 5 και 4. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαδικαστικό. Αύριο το πρωί ψηφίζουμε για την ε, Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Και σήμερα το πρωί βρήκα στο γραφείο μου ένα δώρο, μια σαμπάνια από την πρεσβεία του Βιετνάμ. Και δεν νομίζω ότι είμαι και η μόνη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ θα το επιστρέψω ευγενικά και θα ήθελα να υποδείξω στους συναδέλφους αν και εκείνοι έλαβαν παρόμοιο δώρο, θα πρέπει να αποστείλουμε ένα ε, μήνυμα ότι δεν γίνονται δεκτά τέτοια δώρα πριν από μία τόσο σημαντική ψηφοφορία. Ναι, κάτι τέτοιο είναι ανάρμοστο, λέει ο πρόεδρος. Δεν ε, εντάσσεται στις ε, διπλωματικές προσπάθειες της οποιασδήποτε αντιπροσωπείας, αλλά είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα επηρεαστεί από τέτοια δώρα. Όμως κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για αυρότητα. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι είναι ανάρμοστο να αποστέλλονται δώρα σε επιτροπή που είτε επηρεάζουν είτε όχι, δημιουργούν τον κίνδυνο, έναν κίνδυνο επιρροής, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Εγώ θα φέρω το δικό μου μπουκάλι αύριο το πρωί στην Επιτροπή, για να το επιστρέψω ευγενικά. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Θίξτε σας παρακαλώ το θέμα με το συντονιστές για να αρχίσουμε νωρίτερα. Παράκληση προς τις πολιτικές ομάδες.